Συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ για να ξεκινήσει η συνεδρίασή μας. And let Να σας καλωσορίσω μετά τις θερινές διακοπές. Ελπίζω να περάσετε όλοι πολύ καλά φαντάζομαι η Λιακάδα να σας έδωσε πάρα πολύ ενέργεια για το τελευταίο κοινοβουλευτικό έτος ε, αυτής ε, της θητείας. Ε, Κάρλα, καλώς Η πρότασή μου είναι να περάσουμε στην επίσημη ημερήσια διάταξη. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης χωρίς αλλαγές. Περνάω στις ανακοινώσεις του Προέδρου. Έχουμε διερμηνία σε όλες τις γλώσσες, εκτός από τα αισθανικά και τα αμαλτέζικα. Ελπίζω να μην έχετε πρόβλημα για σήμερα. Η δεύτερη ανακοίνωσή μου είναι πως έχουμε έξι μέλη που ζήτησαν που να συμμετέχουν στο σύστημα της ηλεκτρονικής επιτροπές. Ε, έτσι λοιπόν ε, σημαίνει ότι δεν εκτυπώνονται τα κείμενα για αυτούς τους συναδέλφους, το 8,5% λοιπόν των μελών της Επιτροπής μας. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να σας προσκαλέσω αν σκέφτεστε να συμμετάσχετε κι εσείς, να χρησιμοποιείτε κι εσείς αυτό το σύστημα, το ηλεκτρονικό και να αποφύγετε την εκτύπωση ε, να το δηλώσετε στη γραμματεία. Η τρίτη ανακοίνωσή μου είναι ότι έχουμε ένα νέο συντονιστή από το EFD, ο κ. Τσιμάνσκι. Η επόμενη ανακοίνωση είναι ότι θα έχουμε ένα εργαστήριο στις 18 Σεπτεμβρίου, Τετάρτη, για την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων και των θεραπείων και στις 24 Σεπτεμβρίου θα έχουμε ένα εργαστήριο για την ηλεκτρονική υγεία. Και στις 14 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής μας, θα έχουμε μια δημόσια ακρόαση για τον κανονισμό επισήμων ελέγχων. Τέλος, τελευταία μου ανακοίνωση. Θα έχουμε μία ανταλλαγή απόψεων, ειδική ανταλλαγή απόψεων με τους επιτρόπους Ποτότσινικ και Πίμπαλξ για τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας και θα περιβρίσκεται και ο γενικός, η γενική γραμματέας για τον ειδικό σχεδιασμό, η κυρία Μοχάμετ, και αυτό θα γίνει στις 15 Σεπτεμβρίου από τις 2 και 4 μέχρι τις 5 και 4. Από τον Ιούλιο δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση για συνεχιζόμενους τριμερείς διαλόγους. Αυτές είναι οι ανακοινώσεις που είχα. Και αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, προγραμματισμός του θαλάσσιου χώρου και ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών και θα δώσω το λόγο στον συγητή, τον κύριο Πυρίλο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε στην Ευρώπη το αίτημα της χρήσης του θαλάσσιου χώρου και των παράκτιων ε, ζωνών είναι σε συνεχή αύξηση. Διάφοροι τομείς όπως οι θαλάσσιες μεταφορές, η αλία, η δατοκαλλιέργεια, ο τουρισμός, ε, το, η παραγωγή ε, ενέργειας ε, ζητούν ε, χρήση του θαλασσού χώρου. Έτσι λοιπόν πρέπει να γίνει ένας κατάλληλος συντονισμός χωρίς τον οποίο θα υπήρξε εντατικοποίηση της πίεσης που ασκείται σε πολύτιμους πόρους. Για να απαντήσουμε σε αυτό το σε αυτή την απέτηση η Κομισιόν παρουσίασε το Μάρτιο μια πρόταση οδηγία που δημιουργεί ένα πλαίσιο για το σχεδιασμό του θαλάσσιου χώρου και την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών. Αυτή η απαντά σε μια διαδρομή που είχε ήδη ξεκινήσει από το 2002 με τα κράτη-μέλη που ε, προσχώρησαν στην ε, Σύμβαση της Βαρκελόνης όπου βρίσκουμε πολλούς από τους στόχους που υπάρχουν στην πρόταση η οποία για πρώτη φορά θα αποτελέσει ένα ευρωπαϊκό κανονιστικό μέσο για την ε, κοινή διαχείριση στην ξηρά και στη θάλασσα. Για τη δική μας Επιτροπή πρόκειται για μια σημαντική πρόκληση ε, η αρμόδια επιτροπή ήταν η Επιτροπή Μεταφορών αρχικά, όμως εμείς αποκτήσαμε την αποκλειστική αρμοδιότητα για ορισμένα άρθρα που αφορούν το περιβάλλον και έχουν ένα θεμελιώδη ρόλο για να επιτρέψουν την εφαρμογή και άλλων σημαντικών κανόνων όπως η οδηγία πλαίσιο ε, για το θαλάσσιο χώρο, η οδηγία habitat και η οδηγία για το για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Εγώ ήθελα να ε, αναφερθώ ότι η προστασία του περιβάλλοντος και των παράκτων ζωνών είναι η απαραίτητη προπόθεση για την ανάπτυξη. Αν όλες ε, οι οικονομικές δραστηριότητες ε, που εξαρτούνται από τη θάλασσα ληφθούν υπόψη, βλέπουμε ότι έχουμε μία μπλε οικονομία, μία γαλάζια οικονομία που στην Ευρώπη δίνει 5,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Είναι μία οικονομία που μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλές θέσεις εργασίας, σκεφτούμε όλες τις δραστηριότητες που συνδέονται με τον τουρισμό, τον αηφόρο τουρισμό, τον παράκτη τουρισμό ε, και αυτή η οικονομία θα μπορεί να χρησιμοποιήσει πλήρως το δυναμικό της μόνο αν μπορέσει να προστατεύσει και να διατηρήσει ε, σε καλή οικολογική κατάσταση το θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον. Έτσι λοιπόν η δική μας Επιτροπή πρέπει να ενισχύσει μία ε, η οικοσυστημική προσέγγιση όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 και η ερμηνεία του δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στο να διευκολύνει τη συνύπαρξη μεταξύ των διάφορων δραστηριοτήτων αλλά να δημιουργήσει συνέργειες για να θέσει τις βάσεις για την αηφόρο ανάπτυξη ολόκληρης της επικράτειας. Αυτή η προσέγγιση θα επιτρέψει να εντάξουμε τις οικονομικές, βιολογικές και κοινωνικές πληροφορίες για να φτάσουμε σε μία αποδεκτή ισορροπία μεταξύ της προτεραιότητας, της προστασίας ε, του περιβάλλοντος, της χρήσης των πόρων και ε, των ωφελών για να ενισχύσουμε την αηφόρο διαχείριση και προστασία των διάφορων περιοχών που υπόκειται σε πίεση κλιματικής αλλαγής ε, πρέπει να ακολουθήσουμε μία προληπτική προσέγγιση. Η αρχή της Πρόληψη, πρόληψης ορίζεται στο άρθρο 121 της ε, Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μας επιτρέψει να έχουμε μία αηφόρο ανάπτυξη και να αναπτύξουμε μία στρατηγική διαχείριση του κινδύνου, όχι διορθωτικού τύπου, αλλά που θα βασίζεται σε μία προληπτική δράση σε σχέση με τις ενδυνάμει βλάβες που μπορεί να προκύψουν για το περιβάλλον στην έκθεσή μου έχω δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της διάβρωσης των ακτών. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που δημιουργεί πολύ μεγάλες συνέπειες και για την προστασία της βιοπικιλότητας και για την οικονομική ανάπτυξη και την των ζωνών όλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην εκπόνηση του ε, σχεδίου που ζητάτε από την οδηγία θα πρέπει να ε, προβλέψουμε την προστασία των ε, ακτών, των παράκτηνων ζωνών και επίσης ε, να ε, μπορούμε να αξιολογούμε πώς θα δράσουμε στις περιπτώσεις όπου έχουμε περιοχές που εκτίθενται σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Θα πρέπει να έχουμε μια ορθή διαχείριση του περιβάλλοντος, της θάλασσας αλλά και του παράκτιου περιβάλλοντος. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να καταρτήσουν ένα χάρτη στρατηγικών δραστηριοτήτων μέσω ενός σχεδιασμού με μια αποτελεσματική διαχείριση των πόρων έτσι όπως αναφέρεται στη Στρατηγική Ευρώπη 2020. Στα άρθρα 6 και 7 αναφέρονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να περιλαμβάνονται στα σχέδια διαχείρισης και κατά την άποψή μου πρέπει να προσθέσουμε και ε, τους χώρους για τη δέσμευση και αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακα και πρέπει να αναφερθούμε ε, στο να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για την εξόριξη του αερίου, ε, είτε είναι στην ακτή είτε σε offshore εγκαταστάσεις και πρέπει να σεβόμαστε τις ελάχιστες προϋποθέσεις γιατί κάθε περιοχή έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Θα πρέπει να σεβόμαστε τις εδαφικές ιδιαιτερότητες και να προσέχουμε τις συνέπειες των κλιματικών αλλαγών. Εγώ αυτή την οπτική ήθελα να ενισχύσω στο κείμενό μου την αναγκαιότητα μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ των διάφορων πολιτικών ηθινόντων σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης, ευρωπαϊκό, εθνικό, τοπικό και ταυτόχρονα να εμπλακούν όλοι όσοι έχουν συμφέρον για να προβούν σε, ένα σε μια ολοκληρωμένη διαχείριση ε, όλων των χερσαίων αλλά και θαλάσσιων δραστηριοτήτων. Για πλήρη εφαρμογή της οδηγίας ήθελα να υπογραμμίσω την αναγκαιότητα της ολοκλήρωσης διάφορων εργαλείων συνοχής και του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη θάλασσα θα πρέπει αυτά να διαδραματίσουν ένα κεντρικό ρόλο για την υλοποίηση των στόχων αυτής της οδηγίας. Τώρα θα δώσω το λόγο στους σκιώδη εισηγητές και τους υπόλοιπους συναδέλφους που θα ήθελαν ε, να πάρουν το λόγο για να ακούσουν την απόψή τους. Σας ευχαριστώ. Um, ευχαριστώ κύριε Πυρίλο. Έχω δύο σκιώδεις εισηγητές στον κατάλογό μου που είναι παρόντες και δύο άλλα μέλη της Επιτροπής που θέλουν να πάρουν το λόγο. Να ελέγξω όμως, έχω την κυρία Σνίπερ και την κυρία Κέρλινγκ και την κυρία Λούτσεβα, Τέιβις και Μπονανίνη. Έχουμε άλλον έναν. Περάσατε ωραία το καλοκαίρι, μου φαίνεται. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία Σνίπερ, ε, εκ μέρους του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Πυρίλιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους ε, εισηγητές και σκιώδεις εισηγητές από την Επιτροπή ΤΡΑΝ. Είναι πολύ μεγάλη η σημασία των υδάτων. Ε, νομίζω ότι αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. όχι μόνο επειδή ένα τρίτο των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μένουν ε, εντός 20 χιλιόμετρων από την ακτή. Είναι κάτι που έχει συνέπειες και για πολλούς που ζουν στο εσωτερικό των χωρών και είναι κατανοητό ότι οι ακτές σήμερα αποτελούν και βιομηχανικές ζώνες ε, και ε, χώρο διακοπών ταυτόχρονα. Και είναι ε, και πηγή βιοπικιλότητας, είναι και μέρη για τουρισμό και για αθλητισμό. Και Ε, μπορεί να υπάρχει ε, υπερβολικός φόρτος δραστηριοτήτων ε, στις περιοχές αυτές και θα πρέπει να φροντίσουμε οι παράκτιες αυτές ακτές να μην τις εξαντλήσουμε τελείως. Είναι μια πολλά υποσχόμενη νέα προσέγγιση για να αποφύγουμε κάτι τέτοιο, αυτή η νέα διαχείριση των ακτών και πρόκειται για μια προσέγγιση που βασίζεται ε, σε μια διαδικασία που ε, εγκαίρως ε, εξετάζει τα θέματα αυτά. Και γι' αυτό η οδηγία αυτή θεσπίζει ένα πλαίσιο διαδικασιών και την επικροτούμε. Θα πρέπει να σκεφτούμε επίσης ότι η ίδια η διαδικασία σχεδιασμού και η εξισορρόπηση οικονομικών, οικολογικών και κοινωνικών παραμέτρων θα πρέπει ε, να ε, διατηρηθεί από τα κράτη-μέλη. Κατά τη γνώμη μου, η πρόταση της Κομισιόν ε, υπερβάλλει σε κάποια σημεία και απειλεί την αρχή της επικουρικότητας. Αντί να δημιουργούμε άλλα επίπεδα σχεδιασμού, θα πρέπει να διατηρήσουμε κάποια μέσα και να τα χρησιμοποιήσουμε με πιο ευέλικτο τρόπο και έτσι να έχουμε ε, την ε, μεγαλύτερη δυνατή απόδοση από τους πόρους που έχουμε και ε, να μπορέσουμε να συνδυάσουμε τις διάφορες καλές πρωτοβουλίες και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να υποβάλουμε και κάποιες τροπολογίες που θα οδηγήσουν πιο πέρα τη συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σνίπερ, η Julie Κέρλινγκ από το ECR. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Πυρίλο. Σας ευχαριστώ για την ε, ε, γνωμοδότηση αυτή. Νομίζω ότι εδώ σημαντικό είναι το σημείο κίνησης. Πολλά κράτη-μέλη με ε, μεγάλες ή μικρές παράκτιες ζώνες ήδη έχουν μία σειρά από τα στοιχεία που προτείνονται στο πλαίσιο αυτό. Μερικά έχουν, μερικά δεν έχουν. Ε, πρόκειται λοιπόν για μια κλασική ε, ε, υπόθεση για την Ευρώπη. Η η Κομισιόν τα εξέτασε αυτά. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση στο να έχουμε μια οδηγία πλαίσιο. Να μην ξεχνάμε όμω ότι πρόκειται ακριβώ περί αυτού, περί μια οδηγία πλαίσιο και γι' αυτό θα πρέπει να αποφύγουμε να είναι υπερβολικά αναλυτική, να υπαγορεύει υπερβολικά πολλά πράγματα, διότι σε κράτη-μέλη όπου ήδη υπάρχουν προηγμένα ε, και ε, πολύπλοκα συστήματα, δεν θα πρέπει να χρειαστεί να πρέπει να κάνουν σημαντικές αλλαγές οι οποίες ε, να μην ε, προωθούν ούτε τα περιβαλλοντικά ούτε τα κοινωνικά ζητήματα, αλλά θα επιφέρουν επιπλέον ε, ε, διοικητικό κόστος και και εμπόδια. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε οι βέλτιστες πρακτικές στις χώρες που ήδη χρησιμοποιούν τα περισσότερα από τα μέσα που προτείνονται εδώ ε, θα πρέπει να γίνουν σεβαστά. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ε, όσον αφορά τη διατύπωση στην οδηγία αυτή, ώστε να φροντίσουμε να επιτρέπει ε, αρκετή ευελιξία και να φροντίσουμε να επιτρέπει τον χώρο και χρόνο που απαιτείται για τη συμμετοχή των τοπικών ενδιαφερομένων, διότι όσοι από εμά έχουν ασχοληθεί με ε, τον χωροταξικό σχεδιο, το θαλάσσιο χωροταξικό ε, σχεδιασμό εδώ και καιρό και η δικιά μου περιφέρεια έχει πολύ σημαντική παράκτεια ζώνη, μπορεί, ε, γνωρίζουμε ότι μπορεί κανεί σε μια οδηγία να πει στον κόσμο ότι θα πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ του. Δεν μπορούμε όμω να του υποχρεώσουμε. Μπορούμε να του δώσουμε ένα πλαίσιο συνεργασία και το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να επιτρέπει να, ώστε να αφήνει περιθώριο για τι διάφορε τοπικέ τοπικές ε, προϋποθέσεις. Ε, πρόκειται λοιπόν για... Ε, πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει επικουρικότητα και ο κύριος Πυρίλο όταν μιλάει για τις δραστηριότητες αυτές πρέπει να είμαστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί όσο μιλάμε, όταν μιλάμε για τις εδαφικές δραστηριότητες διότι αυτό αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών. Φυσικά η διαχείριση των ακτών έχει να κάνει με τον σωστό συνδυασμό ε, παράκτιων και ε, ε, χερσαίων δραστηριοτήτων, αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε να μην παραβιάσουμε την κυριαρχία των κρατών μελών, διότι έτσι απλά θα έχουμε διαμαρτυρίες και καθυστερήσεις. Θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες οι οποίες εξετάζουν το θέμα αυτό του θαλάσσιου χωροτοξικού σχεδιασμού από αυτή την οπτική γωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τζούλη, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν μιλώ εκ μέρους ε, της κοιόδους εισηγήτριας ε, Κορίν Λαπάζ που μου έχει ε, υποβάλει κάποιες σημειώσεις από τις οποίες είναι προφανές ότι όχι μόνο στηρίζει τις προτάσεις της Κομισιόν αλλά στηρίζει και την προσέγγιση του κυρίου Μάριο Πυρίλο στην έκθεσή του. Δεν θα εκπλήξει κανέναν ότι η κυρία Λεπάζ στηρίζει μια βιώσιμη προσέγγιση στο, στην ανάπτυξη των, ε, ε της θάλασσας και των ε, παράκτιων ζωνών ε, για την αποφυγή του ανταγωνισμού και την σύγκρουση μεταξύ διαφόρων ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων. Η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει την θαλάσσια οικονομία της, αλλά τονίζει ότι η αρχή της ε, βιώσιμης ανάπτυξης ε, της ε, διατήρησης των πόρων θα πρέπει να αποτελούν ζωτική σημασία κατά το σχεδιασμό της διαχείρισης των ακτών και των παράκτιων διαστηριοτήτων. Επίσης τονίζει αυτό που είπε ο Μάριο ότι έχουμε την αρχή της προφύλαξης και θα πρέπει να προβλέψουμε τα προβλήματα αντί να προσπαθήσουμε να τα λύσουμε μετά εκ των υστέρων. Επίσης ε, χρειαζόμαστε ε, συμμετοχή του κοινού και συνεργασία μεταξύ των διαφορών ενδιαφερομένων. Ε, επιτρέψτε μου να προσθέσω και μια προσωπική παρατήρηση που συμφωνεί με αυτά που είπαν οι δύο τελευταίοι ομιλητέ. Θυμάμαι κατά τη διάρκεια τη πρώτη μου θητεία, νομίζω γύρω στο 2003, Είχαμε την ε, πρώτη έκθεση της Κομισιόν ε, για την ολοκληρωμένη διαχείριση των ε, παρακτήων ζωνών και μπορούμε να σκεφτούμε παραδείγματα από την Ευρώπη όπου υπήρξε παντελής έλλειψη τέτοιας διαχείρισης και είναι δυσάρεστες οι συνέπειες αλλά η αρχή της επικουρικότητας επίσης θα πρέπει να τονιστεί εδώ. Θυμάμαι ότι ήταν πράσινο εισηγητής τότε που ήθελε να γίνει πιο αυστηρή νομοθεσία ε, ώστε η Ευρώπη να γίνει η αρχή διαχείριση για το σύνολο της Ευρώπης, ε, το οποίο είναι ενδιαφέρον διότι τότε ε, ε, συμμετείχε σε εκστρατεία κατά μια συνθήκη που θα, που θα αύξανε τις αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πρόκειται σαφώς για αντίφαση. Λοιπόν, θέλουμε όλοι λογικό σχεδιασμό, θέλουμε βιώσιμες αρχές, αλλά τελικά οι αρμοδιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνουν μόνο μέχρι ένα σημείο και θα πρέπει να τονίσουμε και την αρχή τη επικουρικότητα. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Κρι. Ε, σε ευχαριστώ πολύ που αποτελείς και τη θεσμική μας μνήμη. Ε, αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Κυρία Λιούπτσεβα, εάν ε, έχω προφέρει σωστά το όνομα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα με τη σειρά μου να εκφράσω υποστήριξη για το περιεχόμενο του εγγράφου και την προσέγγιση που επέλεξε ο εισηγητής. Ήρθε ο καιρός πράγματι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει σχετικό έγγραφο. Η οδηγία αυτή συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων νομοθετημάτων που στοχεύουν στην ανάπτυξη των παραθαλάσσιων περιοχών και την στήριξη της διαχείρισής τους να το υποστηρίξουμε το έγγραφο αυτό γιατί με τον τρόπο αυτό θα δείξουμε μια συνεπή στάση απέναντι σε όλα τα θέματα των παράκτιων περιοχών. Είναι σημαντικό το έγγραφο για τα περιβαλλοντικά θέματα που στο κάτω της γραφής είναι η αρμοδιότητά μας. Γιατί, διότι η επέκταση των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, η αύξησή τους κατόγκο είναι γεγονός. Οι πόροι χρησιμοποιούνται εντατικά από την άλλη μεριά, αυτό προκαλεί και προβλήματα. Εκβιομηχάνηση των παραθαλάσσιων περιοχών που προκαλεί πολλές ε, επιπτώσεις ε, στο θαλάσσιο περιβάλλον. Πολλοί άνθρωποι, πολλοί Ευρωπαίοι ζουν στις περιοχές αυτές και οφείλουμε να τους εξασφαλίσουμε καθαρό περιβάλλον και υψηλό επίπεδο ζωής. Έχει λοιπόν μεγάλο ενδιαφέρον το θέμα αυτό για το έργο μας. Ακόμα περισσότερο όταν βρέχονται από την ίδια θάλασσα πλείονες χώρες με διαφορετικά κοινωνικά και πολιτικά συστήματα. Με βεβαίως όλα όσα συνεπάγεται η έντονη κυκλοφορία και η βιομηχανική δραστηριότητα. Αυτά συχνά έχουν ως συνέπεια την ρήπανση των νερών, την ρήπανση των εδαφών, των παραθαλάσσιων περιοχών. Η οδηγία λοιπόν δεν θεωρώ ότι παραβιάζει τις εξουσίες των χωρών σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση των θεμάτων των παραθαλάσσιων περιοχών τους. Αυτά διατηρούν την κυριαρχία, αλλά συμβάλλει στην θεμελίωση μιας συνεργασίας όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει μια πλατφόρμα για τον συντονισμό των διαφόρων δραστηριοτήτων χωροτακτικών και άλλων. Δεύτερο, επίσης όμως σημαντικό, οι προστατευόμενες περιοχές της Natura 2000 θα πρέπει να περιληφθούν. Και αυτό θα είναι μια σημαντική συμβολή της ε, παρούσας οδηγίας. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κύριε Λίψεβα. Ο κύριος Χρυσόγελος, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την πρότασή της και τον εισηγητή για την έκθεσή του. Ε, τον Οκτώβριο του 2012 οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Θαλασσίων Υποθέσεων υιοθέτησαν τη διακήρυξη Λεμεσού με στόχο να προωθήσουν ένα ισχυρό θαλάσσιο πυλώνα για να στηρίξουν τη στρατηγική Ευρώπη 2020. Η Κομισιόν υποστηρίζει ότι η γαλάζια οικονομία προσφέρει ευκαιρίε για βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση. Η γαλάζια οικονομία, η οικονομία δηλαδή που βασίζεται στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον, μπορεί πράγματι να συμβάλλει τα μέγιστα στην κοινωνική ευημερία, τη δημιουργία θέσεων εργασία και στην έξοδο από την κρίση. Απ' την άλλη όμω η αυξανόμενη παρέμβαση στη θάλασσα και σε ακτέ μπορεί να θέσει σε κίνδυνο αυτά τα ίδια τα αγαθά. Ήδη υπάρχει μεγάλη χρήση των ακτών και τη θάλασσα, Τεράστιε συγκρούσει εντοπίζει στα χωρικά ύδατα, αλλά και πέρα από αυτά, χωρί να υπάρχει κατάλληλη διαβούλευση ή περισσότερο θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και σχέδια ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτα ζώνη. Για να αντιμετωπιστούν οι αυξανόμενοι χρήση των παράκτων και θαλάσσιων περιοχών, οι συνέπειε κλιματική αλλαγή, οι κίνδυνοι από τη διέλευση πετρελαιοφόρων ή πλοίων με χημικά, η διάβρωση, η φυσική κίνδυνη, η μετατροπή της θάλασσα σε οικόπεδα με αποκλειστική χρήση στην εξόρυξη πετρελαίου, φυσικού αερίου ή μεταλλευμάτων, πρέπει να μειωθούν οι πιέσεις στην ευαίσθητη αυτή ζώνη μέσω ολοκληρωμένη, συνεκτική και συνετής διαχείρισης. Ενώ πολλέ χώρε χρειάζεται να επιταχύνουν το χωροταξικό σχεδιασμό στην ξηρά, είναι επίση ανάγκη ο χωροταξικό σχεδιασμό να προχωρήσει γρήγορα και στη θάλασσα και στην παράκτια ζώνη, πριν οι λάθο πρακτικέ στην ξηρά επεκταθούν πλήρω σε αυτέ τι ιδιαίτερα ευαίσθητε περιοχέ χρειαζόμαστε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα πλαίσιο για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που θα περιλαμβάνει και την παράκτια ζώνη και θα συνδυάζεται με αυτόν για την ξηρά, μέσω ενό ολοκληρωμένου δηλαδή χωροταξικού σχεδιασμού ξηρά και όπου υπάρχει ακτή και θάλασσα. Είναι σημαντικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό να λειτουργεί συνεκτικά σε περιφερειακό, εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο, μια και τα θαλάσσια οικοστήματα δεν περιορίζονται στα εθνικά ή διοικητικά σύνορα. Δεν είναι φυσικά κάτι εύκολο. Απαιτεί καλό συντονισμό, διάθεση επίλυση προβλημάτων. Για παράδειγμα, υπάρχουν συνοριακέ διαφορέ ή ασαφεί σύνορα, αντιτιθέμενε δραστηριότητε και διαφορετικά συμφέροντα. Χρειάζεται όμω κοινή μεθοδολογία, συγκέντρωση και επεξεργασία αξιόπιστων δεδομένων, συμμετοχή στη διαβούλευση των διαφορετικών κοινωνικών εταίρων. Υπάρχουν ορισμένε καλέ προσπάθειε σε περιφερειακό ή σε διασυνοριακό επίπεδο, για παράδειγμα μεταξύ Γερμανία και Πολωνία, σχέδια στην περιοχή του Ατλαντικού ή τη Βαλτική, αλλά και στο πλαίσιο του Μεσογειακού Σχέδιου Δράση του Προγράμματο ΕΕ για το Περιβάλλον, UNEP-MAP, κυρίω στο πλαίσιο εφαρμογή του Πρωτοκόλλου για την Παράκτια Ζώνη. Η εφαρμογή του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού στι τρει μακροπεριφέρειε Μεσογείου θα μπορούσε να βοηθήσει την πρόθεση κοινών διασυνοριακών πιλωτικών πρωτοβουλειών σε μια περιοχή όπου ο χωροταξικό σχεδιασμό δεν έχει προχωρήσει ακόμα ικανοποιητικά. Όμω, επιμέρου και συχνά αποσυμματικέ ή χωρί συνέχεια πρωτοβουλίε δεν θα φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα Πολλά κράτη-μέλη έχουν καθυστερήσει υπερβολικά τον χωροταξικό σχεδιασμό στην ξηρά. Είναι πιθανόν λοιπόν να καθυστερήσουν ακόμα περισσότερο το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ενώ οι εξελίξει και οι παρεμβάσει σε αυτό το χώρο είναι ήδη πολύ έντονε. Εξορίξει, άντλη πετρελαίου και φυσικού αερίου, ανεξέλεγκτη χάραξη θαλάσσιων διαδρομών, πετρελοφόρων και άλλων σκαφών με επικίνδυνα φορτία, μέσα ή κοντά σε ευαίσθητε οικολογικέ περιοχέ, εκτεταμένα δίκτυα αγωγών πετρελαίου, ηλεκτρικών χαλωδίων χωρί να έχει προηγηθεί ένα πραγματικό σχεδιασμό και να έχουν συμφωνηθεί οι χρήσει θαλάσσιε περιοχέ. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία τη Κομισιόν για μια ευρωπαϊκή οδηγία που θέτει ένα κοινό πλαίσιο για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτια ζώνη που μέχρι τώρα ήταν σε επίπεδο θελοντικών πρωτοβουλειών. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός χρειάζεται να βασίζεται σε κοινέ για όλους κατευθύνσει και κοινά standards, αλλιώς θα υπάρξει σύγχυση, διαφορετικές προσεγγίσεις αναποτελεσματικότητα, ενώ την ίδια στιγμή θα ενισχυθεί η καταστροφική εκμετάλλευση θαλάσσιων και παράκτων πόρων. Μερικά σημεία. Τα θαλάσσια και παράκτα οικοστήματα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα. Απαιτεί λοιπόν να ακολουθεί η προσέγγιση του οικοστήματο ω εργαλείο για το σχεδιασμό και να λαμβάνονται υπόψη υπηρεσίε που προσφέρουν τα οικοστήματα αυτά. Η αρχή τη πρόληψη έχει ιδιαίτερη σημασία και στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Η υπευθυνότητα διαμορφώνεται μέσα από τη συμμετοχή και τη διαβούλευση. Τα σχέδια αυτά σε περιφερειακό, εθνικό και δεσμευτικό επίπεδο πρέπει να διαμορφωθούν μέσω από εκτενή διαβούλευση με τι περιφερειακέ και τοπικέ αρχέ, του πολίτε και την κοινωνία των πολιτών. Τα σχέδια είναι αναγκαίο να διασφαλίσουν, να διασφαλίσουν τόσο την κοινωνική συνέχεια. <laughs> Παρακαλώ ολοκληρώστε, παρακαλώ ολοκληρώστε. Uh, welcome, Mrs. Stutzer, Uh, your first Καλώς ήρθατε και εσείς κυρία Φιούτσα, είναι και η πρώτη σας ε, παρέμβαση στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η ολοκληρωμένη διαχείριση των παραθαλάσσιων περιοχών είναι σημαντική υπόθεση. Νομίζω επίσης ότι είναι τόσο σημαντική που να άπτεται της επιβίωση του πλανήτη μας. Είμαι από την Κροατία. Γνωρίζετε ότι η Αδριατική θάλασσα είναι μια θάλασσα που βρέχει και τις δικές μας ακτές καθώς και τις ακτές άλλων χωρών. Έχουμε μια προστατευμένη οικονομική ζώνη, αλλά αυτό είναι άλλη υπόθεση. Βρέχει η θάλασσα αυτή λοιπόν χώρες με διαφορετικό βαθμό οικονομικής ανάπτυξης και που χειρίζονται τα της θάλασσας με διαφορετικούς τρόπους. Χρειάζεται λοιπόν να εξασφαλιστεί μια ισορροπία ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και της, και της οικονομίας χωρίς ωστόσο να θίξουμε την αρχή της επικουρικότητας Χρειαζόμαστε την οδηγία για να μπορέσουμε να εξισορροπήσουμε έτσι την ε, προσέγγιση μας αυτή, τους κανόνες που θα εφαρμόσουμε. Γι' αυτό και πρέπει να ψηφιστεί η οδηγία για να δοθεί στις χώρες μέλη και ένα περιθώριο διαχείρισης. Να μην θυγεί η κυριαρχία τους δηλαδή. Έχοντας υπόψη Μη λησμονώντας τι έλεγαν και οι, οι της Αμερικής ότι δανειστήκαμε την γη αυτή από τα παιδιά μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν ε, θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Περίλο για την έκθεσή του που την υποστηρίζω απόλυτα και για σημαντική δουλειά εμπλουτισμού μιας οδηγίας που είναι ήδη πολύ σημαντική όπως αυτή που πρόσφατα παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για, το, για τον προγραμματισμό του θελασσίου χώρου κληροκυρωμένου διαχείριση των πράκτων ζωνών. Πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα. Η οδηγία είναι ιδιαίτερα σκόπιμη μία ε, ορθή, ένας ορθός προγραμματισμός ε, του θελασσίου χώρου και μια ολοκληρωμένη διαχείριση των πράκτηρων ζωνών είναι κάτι απαραίτητο για την αηφόρο ε, ανάπτυξη της επικράτειας ε, και γι' αυτό χρειαζόμαστε συντονισμένα και λεπτομερή σχέδια. Επίσης είναι σημαντικό να προβλέπουμε πώς θα λαμβάνουν υπόψη τα σχέδια αυτά και την οδηγία για τον περιβαλλοντικό ακτιτυπό. Θα ήθελα βέβαια να παρουσιάσω ορισμένα σχόλια, ορισμένες πτυχές στο συνάδελφο που θα έπρεπε να τονιστούν περισσότερο. Η κατάσταση των υδάτων πρέπει να υπάρχει μια πραγματικά ολοκληρωμένη διαχείριση του θαλάσσιου χώρου και με συγκεκριμένη παρεμβολή στις δραστηριότητες πρέπει να ληφθούν υπόψη στον καθορισμό των σχεδίων του άρθρου 7 και στην κατάσταση που συναντάμε σε ό,τι αφορά ε, τις αποθέσεις της χωματερές και επίσης ε, πρέπει να έχουμε και κατάλληλα συστήματα βιολογικού καθαρισμού. Αυτό αποτελεί κάτι πολύ σημαντικό για την επικράτεια, ίσως για να μπορεί να καταναλώνεται ε, και το νερό και να χρησιμοποιείται για τη γεωργία. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ε, θαλάσσιες διαδρομές, νομίζω ότι πρέπει να ε, αναφερθούμε περισσότερο στο στόχο της ασφάλειας των οικοσυστημάτων όπως και στην ασφάλεια των μεταφορών. Η σχέση που υπάρχει μεταξύ των διαδρομών, ε, των θαλάσσιων διαδρομών αλλά και ε, των θαλάσσιων ε, ζωνών είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έχουμε δει τι συμβαίνει στη Βενετία και τι συνέβη και στα ύδατα της Τοσκάνης. Όλα αυτά κρούν τον κόδυνα του κινδύνου για το μέλλον. Οι διαδρομές χιλιάδων σκαφών ε, που μεταφέρουν τοξικά φορτία και επικίνδυνα φορτία μπορεί να αποτελούν απειλές για το οικοσύστημα και ε, είδαμε και στο πρόσφατο παρελθόν ότι ένα τέτοιο ναυάγιο οδήγησε σε ε, ιδιαίτερες βλάβες του οικοσυστήματος και οι κίνδυνοι αυτοί είναι πάρα πολύ προφανείς, επομένως πρέπει τα σχέδια διαχείρισης να λαμβάνουν υπόψη και το σχεδιασμό των θαλάσσιων διαδρομών των πλοίων. Γιατί αν έχουμε βλάβη του οικοσυστήματος, τότε ακυρώνουμε οποιαδήποτε μορφή ανάπτυξης, ακόμη και τουριστική. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο σύντομα παρακαλώ στην Κομισιόν, η κυρία Ευχαριστώ και καλημέρα σε όλες και όλους. Ολίγα σχόλια για την οδηγία, καθώς και απαντήσεις σε παρατηρήσεις δικές σας, αφού πρώτα ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεσή του. Θα επανέλθω όμως σε λίγο και ευχαριστώ βεβαίως και όλες και όλους τους ομιλητές. Υπενθυμίζω ότι η οδηγία αυτή για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτων περιοχών εντάσσεται στην προσπάθεια της Κομισιόν να αναπτύξει την γαλάζια οικονομία και γαλάζια ανάπτυξη και επομένως εκεί αντιμετωπίζονται ορισμένες συγκεκριμένες προκλήσεις τις οποίες θα ήθελα να τονίσω. Για την ώρα δεν υπάρχει συντονισμός της διαχείρισης θαλάσσιων και παραθαλάσσιων περιοχών με αποτέλεσμα ανταγωνισμό για την χρήση τους, ανεπαρκή προστασία των θαλάσσιων πόρων, αβεβαιότητα και έλλειψη προβλεψιμότητας για την πρόσβαση στον θαλάσσιο και παραθαλάσσιο χώρο, το οποίο βεβαίως δεν εξασφαλίζει το βέλτιστο δυνατό επιχειρηματικό κλίμα. Και σε ό,τι αφορά το περιβάλλον το οποίο ιδίω μας απασχολεί, αυτό αντιμετωπίζει σημαντικές πιέσεις το θαλάσσιο περιβάλλον δηλαδή, που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο ζωτικούς πόρους στους οποίους βασίζεται η οικονομία μας και γι' αυτό χρειάζεται να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή. Υπενθυμίζω ότι υπάρχουν αυξημένες απαιτήσει αλλά και ευκαιρίες βεβαίως που προκύπτουν από κοινοτικέ πολιτικές είτε πρόκειται για αλληλεία, για ε, πολιτική προστασία του περιβάλλοντος, ενέργεια κλπ. Όπως είπατε ορισμένοι εξημών πρέπει να συντονιστούν οι δραστηριότητες αυτές, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουμε την αποτελεσματικότητά τους και να επιτύχουμε έτσι και οικονομικούς και περιβαλλοντικούς στόχους. Αυτός ο συντονισμός είναι ο στόχος της παρούσας οδηγίας. Τα προβλήματα τώρα που έχω εντοπίσει και βεβαίως δεν μπορούν να επιληθούν μοναχά με τούτην εδώ την πρόταση, ούτε άλλωστε έχει αυτό το σκοπό. Πολλοί και πολλές από εσά τονίσατε ότι υπάρχει ανάγκη οι εθνικές αρχές να πράξουν τα δέοντα. Εμείς ήδη επεξεργαζόμαστε ορισμένα θέματα. Η δική μας συμβολή με την παρούσα πρόταση έχει στόχο να συμπληρώσει τις δραστηριότητες των χωρών μελών. Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος αλλά και ε, Θαλάσσιων θεμάτων έχουμε αναλάβει την εργασία αυτή και θέλουμε να συνεργαστούμε με τις εθνικές διοικήσεις των χωρών μελών. Αυτό είναι σημαντικό θέμα και το τονίζω λοιπόν για μια ακόμη φορά. Θα ήθελα επίσης να τονίσω και το θέμα της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που έχουν ληφθεί υπόψη στην πρόταση. Πρόκειται για οδηγία πλαίσιο η οποία προβλέπει διαδικαστικές ρυθμίσεις που θα πρέπει να γίνουν σεβαστές, αλλά σε ό,τι αφορά το ουσιαστικό περιεχόμενο των μέτρων καθώς και τον χρονισμό τους, αφήνει μεγάλη ευκαμψία στις χώρες μέλη έτσι ώστε να ρυθμίσουν τα πράγματα αυτά στο εθνικό και περιφερειακό επίπεδο κατά το δοκούν. Αποσκοπούμε στην αύξηση της, στη, μάλλον στην ανάπτυξη στην εξασφάλιση της ανάπτυξης, στην προστασία των πόρων, να παραμείνουν αυτοί βιώσιμοι και νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό πρέπει να συντονιστούν όλες οι σχετικές πολιτικές. Ένα άλλο ε, θέμα που είναι σημαντικό για μας είναι ο διαμεθοριακός χαρακτήρας. Είναι σημαντικό οι δραστηριότητες μεταξύ των χωρών μελών να συντονίζονται, διότι γνωρίζουμε ότι οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα είναι συνήθως διαμεθοριακές. Επανέρχομαι τώρα στην έκθεση, σύντομα. Όπως είπα, μας ικανοποιεί ιδιαίτερως η πρόταση του εισηγητού, που νομίζουμε ότι στηρίζει την προσέγγιση της Κομισιόν και περιλαμβάνει χρήσιμες συστάσεις για την νομοθετική διαδικασία. Για παράδειγμα, αναφέρει το θέμα της διάβρωσης των παραθαλάσσιων ε, περιοχών και άλλα σχετικά. Ένα συγκεκριμένο θέμα που ανέφερε ο εισηγητής σχετικά με τις δραστηριότητες για την αποθήκευση, μάλλον δέσμευση και αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα, καθώς επίσης την εξόρυξη σχιστολιθικού αερίου κλπ. Αυτά βεβαίως μας βρίσκουν ανοιχτούς για συζήτηση. Γιατί να περιληφθούν δηλαδή στην οδηγία θεωρούμε ότι πολλές από τις προτάσεις που γίνονται στην έκθεση με κάποιο τρόπο μπορεί να περιληφθούν στην πρόταση οδηγίας, ίσως όχι με τόσο ορατό τρόπο, αλλά πάντως θα το επανεξετάσουμε και θα δούμε πώς θα τα καλύψουμε ενδεχομένως και στην αιτιολογική έκθεση. Συμπεραίνοντας, θα μελετήσουμε την έκθεση σας ακόμη περισσότερο, όπως και τις προτάσεις των σκιωδών εισηγητών. Έχουμε και ερωτήσεις που αποζητούν περαιτέρω διευκρίνηση και θα προχωρήσουμε. Παρακαλούμε πάντως την Επιτροπή σας να προχωρήσει γρήγορα στην συζήτηση, ώστε οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο να μπορέσουν να αρχίσουν το δυνατόν σύντομότερο. Διότι, εάν μπορέσει η συμφωνία να ε, συναυθεί σύντομα μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Αυτό θα είναι προς όφελος όλων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία μου. Φτάσαμε στο τέλος της συζητήσεως. Κύριε Σιγητά, επιθυμείτε να λάβετε πάλι το λόγο. Ναι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο και την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους ε, που εκτίμησαν τη δουλειά μου. Ανέκυψαν κάποιες αποχρώσεις ε, που σίγουρα θα πρέπει να τις λάβουμε υπόψη και να καταλήξουμε στη βαλτιστή δυνατή λύση, γιατί και εγώ θεωρώ πως αυτή η οδηγία πλαίσιο είναι σημαντική και μάλιστα το ανέφερε και ο Κρίς Ντέιβις κατά κάποιο τρόπο. Τα κράτη-μέλη πρέπει να κατανοήσουν ότι ο θαλάσσιος χώρος και η διαχείριση των παράκτων ζωνών είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να εξεταστεί και σε εσωτερικό επίπεδο, αλλά θα πρέπει να ειδωθεί και συνολικότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ πολύ. προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 12 Σεπτεμβρίου στις 12 στην Επιτροπή ΕΝΒΗ. Θα ψηφίσουμε στις 17 Οκτωβρίου. Η Τραν στις 5 Νοεμβρίου θα ψηφίσει και στην Ολομέλεια τον Δεκέμβριο. Έτσι, ολοκληρώσαμε τη συζήτηση για το σημείο 3 της ημερησίας διάταξης και μπορούμε να προχωρήσουμε στο σημείο 4 της ημερησίας διάταξης. Ε, θα ήμουν πολύ ικανοποιημένος αν είχα τώρα κατάλογο των ψηφοφοριών. Έχουμε την έκθεση ΧΑΟΚ Ξεκινάμε κατευθείαν. Η εισηγήτρια θέλει κάτι να πει. Πολύ σύντομα. Δεν θα αναφερθώ στις αρχές μου. Η αρχή μου είναι να, μην, ε, είναι να επανέλθουμε στο ε, σχέδιο προϋπολογισμού. Ε, θα ήθελα μόνο να πω ότι το Προεδρείο μας από το Προεδρείο μας λείπει κάποιος όταν συζητάμε για τον προϋπολογισμό. Συνήθως ε, είναι η Εμίλια παρούσα. Ε, γιατί δεν είναι η Εμίλια εδώ, διότι παντρεύεται. Συγχαρητήρια λοιπόν, τις ευχόμαστε. Και εύχομαι μετά το γάμο να συνεχίσει να είναι εξίσου ευτυχισμένη. Μπορούμε να ψηφίσουμε. Ωραία, ε, ακούσαμε λοιπόν μια ευχάριστη δήλωση της Utah Hawk και από εμά ευχές προς την Εμίλια και Προχωράμε στην ε, ψηφοφορία. Τροπολογία 6328. Ε, Έχετε όλοι έτοιμες τις κάρτες σας. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6303. Ζανώνη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6338. Υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. 63-34 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 63-21 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 63-35 υπέρ, 63-35 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 63-22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 63-23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 63-24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 63-12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Το ελέγξουμε. Αρχή της ψηφοφορίας. 63-12. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 63-26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 63-25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 63-06 και 63-42 οι νόμιες υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 63-07 και 63-40 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. 6341, 6308 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 6309 και 6339 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 6310 υπέρ, κατά, αποχές, δεν είναι πολύ σαφές, ε, ελέγχουμε ηλεκτρονικά 6310. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 63-13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 63-02 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 63-16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 63-17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 63-01 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 6301, ε, αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 6318 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6319 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6320 υπέρ κατά απόχεια εγκρίνεται. 63-45 καταπίπτει. 63-47 υπέρ. Κατά. αποχες συγκρινεται εγκρίνεται. 63-46 υπέρ. Κατά. αποχες απόχεια εγκρίνεται. 63-48 υπέρ. Κατά. απόχεια εγκρίνεται. 63-00 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 6304 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 6311 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 6314 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 6337 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 6336 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 63-05 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 63-27 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 63-15 υπέρ, κατά, αποχές δεν είναι πολύ σαφές. Ελέγχουμε. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 63-49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ελέγχουμε. Ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 63-29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 63-30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται με την πλειοψηφία. 63-31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 63-32 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. 63-44 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει η 63-33 και ολοκληρώσαμε αυτό το σημείο και προχωράμε στην γνωμοδότηση. Ε, εδώ έχουμε μονοψήφιες τροπολογίες. Ε, τροπολογία 1, το πρώτο μέρος. Ε, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος υπέρ, κατά, αποχές. Δεν είναι σαφές. Ελέγχουμε το δεύτερο μέρος ηλεκτρονικά. Τροπολογία 1. Δεύτερο μέρος ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Πρώτο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές ε, δεν είναι σαφές. Ε, ελέγχουμε το δεύτερο μέρος της τροπολογίας 3. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Με ε, προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ κατά, αποχές δεν είναι σαφές, ε, ελέγχουμε την 7 ηλεκτρονικά, αρχή της ψηφοφορίας, ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Τροπολογία 8, υπέρ, κατά, αποχές επίσης εγκρίνεται. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 8. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορία. Εγκρίνεται με την ίδια πλειοψηφία. Προχωράμε στην τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την ε, γνωμοδότη... τη γνωμοδότηση όπως τροποποιήθηκε. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορία. 43 υπέρ, 4 κατά, 3 αποχές. Συγχαρητήρια στη Γιούτα Χάουκ. Έχουμε προφορική ερώτηση η κατάσταση της Ευρωπαϊκής Αγοράς Άνθρακα το 2012. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την ε, γνωμοδότηση αυτή, αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ομόφωνα. και ψηφίζουμε ένα διορθωτικό για τις σοβαρές διασυνοριακές απειλές για την υγεία. Ο Ζήλ Παρνιό θέλει κάτι να πει. Όχι, είναι αυτονόητο το θέμα. Υπέρ. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ, λήξη της ψηφοφορίας. 48 <clears throat> υπέρ, κανείς κατά καμία αποχή, εγκρίνεται το διορθωτικό. Η επόμενη συνεδρία θα πραγματοποιηθεί στις 18 Σεπτεμβρίου, 9 η ώρα, μέχρι τις 12.30 και μετά από τις 3 μέχρι τις 6.30 το απόγευμα. Στις 10.30 θα συνεδριάσουν οι συντονιστές. Εύχομαι λοιπόν καλό μεσημέρι σε όλους τους υπόλοιπους και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο.